So dear colleagues, please Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος. Ας καλωσορίσουμε τον Έλκε Κιόνιχ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ενίου Συμβουλίου Εξυγένσης. Είναι μεγάλη μας χαρά. Θα σε έχουμε κοντά μας την πρώτη σας εμφάνιση φέτος, αλλά και για πρώτη φορά από την ανανέωση της εντολής σας. Άρα με μεγάλη χαρά σας ξεκινήσουμε έναν καινούργιο κύκλο συνεργασίας και στενής θεσμικής συνεργασίας. Τα είχαμε πει τελευταία φορά τον Δεκέμβριο, οπότε και ψηφίσαμε για την ανανέωση της εντολής σας, υπέρ της ανανέωσης εντολής σας, ενώ ώψη και των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί. Έχουμε τώρα τον κύριο Γιάσπερ, καινούργιο μέλος του Δικαίου Συμβουλίου της ε, Κεντρικής Τράπεζας και του και μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με την ε, Λετωνία για τη σχετική απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας οπότε Έχουμε και τώρα κάποια άλλα θέματα σε σχέση με την Banco Popular. Και σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο Κοινοβούλιο και θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια για τα όσα έχουν συμβεί στις περιπτώσεις εκείνες. Έχουμε επίσης και κάποια νέα μέτρα στα πλαίσια της δέσμης τραπεζικών ε, νομοθετημάτων. Άρα το μενού είναι πλούσιο για την ανταλλαγή απόψεων και σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πολύ μου αρέσει που βρίσκομαι ενώπιον της Επιτροπής σας γιατί πρόκειται κάτι το αξιόλογο. Ε, εκπροσωπείτε τους πολίτες για μας εδώ είναι πολύ σπουδαίο. Οπότε, όπως και εσείς αναφέρατε, το μήνυμα είναι πάρα πολύ πλούσιο και η συζήτηση θα πρέπει να είναι ειλικρινής. Όπως είπατε και εσείς, ο κύριος Γιάσμπεκ, χθες έτυχε της ε, επικύρωση της εντολής του από το Συμβούλιο. Θα τα συζητήσουμε σύντομα. Θα έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μόλις είναι έτοιμος και έτσι θα είναι πλήρες το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, θα πρέπει να πούμε δύο λόγια και για την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, δύο γιατί ήδη αναφέρατε για κάποια έγγραφα που έχουν σχέση με τα της εκαθάρισης και εξυγίανσης της Banco Popular. Επίσης αναφέρατε και τα της τράπεζας ABLV ε, και θα έχουν να ε, ε, ανταλλάξουν κάποιες απόψεις για την οδηγία εξυγίανσης, τον κανονισμό CRR και το CRD, ο οποίο όλων αυτών έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Αλλά πρώτα-πρώτα, όσον αφορά τις συστάσεις και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, τον Νοέμβριο δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα του 18, ήδη τα συζητήσαμε το Δεκέμβριο. Άρα εδώ να μην σταθούμε. Όμως δύο μήνες αφού δημοσιοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα, το ελληνικό συνεδρίο έδωσε στη κάποιες ε, συστάσεις που απορρέουν από τον οικονομικό έλεγχο του δευτέρου εξαμήνου του 16 αρχών του 17. Και άρα πριν τον πραγματισμό του 17 όλα αυτά αποκρισταλώνονται. Εμεί θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ θετικές αυτές οι συστάσεις και θα τις αξιολογήσουμε επίσης. Έχουμε τις ε, συστάσεις του 17 και έχουμε επίσης το πολιτέ, πρόγραμμα οπότε υπάρχουν πολλές αντιστοιχίες για να πούμε την αλήθεια Φερρυπίν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, τον προσωπικό υπήρχε ένα ποστό επικρίσεων στην έκθεση, αλλά τώρα έχουμε καινούριο πρόγραμμα 300 στο προσωπικό και θα έχουμε εξαρτηθεί πλήρως αυτό το πρόγραμμα για τους ανθρώπινους το Τέλος το τους επίσης ήταν και το θέμα του MRL και σχετική μας πολιτική για τις αποφάσεις τις φετινές αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτό το μέτωπο γιατί το 2018 θα πρέπει για όλους τους τραπεζικούς ομίλους και σημαντικά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε, αυτές τις, ε, σε αυτές, ε, τους τραπεζικούς ομίλους θα πρέπει να καθοριστούν αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις. Οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα κάνουμε κάτι όσον αφορά το, τα, τα, τα εμπόδια στο ε, αξιόχρεο και θα πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί συμφωνίες της συνεργασίας με τις Εθνικές Αρχές Εξυγίανσης. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα επικαιροποιήσουμε τα όσα ισχύουν όσον αφορά την εξυγίανση και όλα αυτά θα μας απασχολούν στο δεύτερο εξάμεινο του 2018 οπότε και θα επικοιροποιήσουμε επίσης βαθμιαία τις σχετικές διατάξεις. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς όλες οι τράπεζα συμμορφωθούν μετά τις εξυγίανσεις ε, μέχρι το 2020 που λύγει η θητεία μας. εμεί θεωρούμε ότι τα πράγματα προχωράνε αργά, λένε ότι είναι γρήγορα. Ε, πάντως προς το παρόν κανείς τραπεζίτης που είναι υπεύθυνος δεν θα πρέπει να περιμένει τις ε, αποφάσεις του Συμβουλίου Εξυγένσης. Θα πρέπει επομένω να άρουμε όλα τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν, γιατί το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει λόγος αναμονής. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και στέλνουμε σε εγώ στις τράπεζες, εγώ και οι συνάδελφοι. Θέλουμε αυτό να αποδοσκαρπιστώ Τώρα και να δούμε την πρόσφατη ε, απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια όσον αφορά την ε, έκθεση που αφορά την εξυγίανση της ε, Banco Popular. Αρχές Φεβρουαρίου είχαμε την ε, διαβούλευση, πήρε χρόνο, οπότε δημοσιεύτηκαν σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεση. Η λεγόμενη αξιολόγηση του 2 ε, και το σχέδιο εξυγένσης του 16. Θα πρέπει βέβαια ακόμα να θεωρήσουμε απόρριτα κάποια κομμάτια αυτής της ε, διαδρομής. Και γιατί αφορά την Ευρωπαϊκή Κίτρα Τράπεζα ή επειδή αφορά κάποιους εμπορικά συμφέροντα της ε, Banco Popular. Οπότε για αυτό πρέπει να πούμε ότι το Συμβούλιο Εξηγένσης θα πρέπει να σεβαστεί την ε, ανεξαρτησία του αξιολογητή. Χρειάζεται κάποιο χρόνο φτιάξει όλους και όπως και εσείς ανυπόμονα περιμένουμε την τρίτη ε, αξιολόγηση και έχουμε σχεδίσει τον αξιολογητή ότι περιμένουμε πώς και πώς, ε, όσο δηλαδή νωρίτερα να ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο στάδιο, αλλά από αυτούς εξαρτάται μια που είναι όργανο ανεξάρτητο κανείς, δεν θα ήθελε να κατηγορηθεί ότι πίεσε τους αξιολογητές γιατί πρέπει να τους αφήνουμε κάποιο περιθωρισμό. Τώρα για να δούμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με το Φεβρουάριο ε, για την ε, Λετωνική Τράπεζα και την ε, θηγατρική της στο Λουξεμβούργο. Αυτές οι τράπεζες βρέθηκαν υπό εκαθάριση. Ε, η πτώχευση, η εκαθάριση μάλλον διέπεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου, είναι ιδιότυπη αυτή η υπόθεση, οπότε θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε, γιατί πρώτα-πρώτα μας υπενθυμίζει, μας θυμίζει μάλλον αυτή η υπόθεση έντονα ε, το, το γεγονός ότι η πτώχευση παραμένει μονόδρομος για πολλές τράπεζες. Οπότε και το Συμβούλιο Εξυγίανσης αναλαμβάνει τα ενία. Και το σχέδιο της εξυγίανσης του 2017 ήδη είχε δείξει ότι υπήρχαν προβλήματα σε σημαντικές λειτουργίες των κρατών μελών, όπως επίσης και το ότι δεν υπήρχε έντονο ε, κρατικό συμφέρον και επομένως η προτιμητέα στρατηγική θα ήταν η πτώκευση. Αλλά επίσης ανέδειξε αυτή η υπόθεση κάτι άλλο. Το πόσο σημαντικό θέμα είναι η εναρμόνιση του πτωχευτικού δικαίου των τραπεζών. Γιατί ο μηχανισμός εξυγίανσης πρέπει να καλύψει 19 ή περισσότερες διαφορετικές ε, διαδικασίες πτώχευσης. Οπότε η αξιολόγηση failing or likely to fail δεν ε, οδηγεί αυτόματα, δεν είναι δεδομένο ότι οδηγεί σε κάποια κριτήρια πτώχευσης και καθάρισης. Οπότε γενικά μπορούμε να πούμε, και όχι μόνο σε αυτήν την περίπτωση, ότι θα πρέπει έτσι να αποκλείσουμε κάποιο είδους επιλήψιμα κίνητρα. θα πρέπει η κατάληξη να είναι ίδια για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει η κατάληξη της πτωχής διαδικασίας να εξαρτάται από τις διαφορές των εθνικών πτωχευτικών δικαίων. Οπότε, θα πρέπει ο ενιαίος μηχανικός εξυγίανσης να ξεκαθαριστεί στο πώς εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Και θα πρέπει επίσης να δούμε στο αν ε, κάποια υπόθεση, κάποια περίπτωση θα οδηγηθεί σε εξυγένση ή σε πτώχευση δυνάμει του εθνικού δικαίου. Άρα θέλουμε εναρμονισμένο σύστημα το οποίο αφορά τους νομοθέτες. Και λέγοντας νομοθέτες ενώ εσάς. Εσείς μπορείτε να το κάνετε μόνο αυτό οπότε για να καταλήψουμε κάπου τώρα αναδείτε το θέμα της δέσμης τραπεζικών μέτρων. Και παρακολουθούμε από πλευρά Συμβουλίου Εξυγένση την προβληματική εδώ στην ε, Επιτροπή σας και βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο συνεχώς ε, ανακύπτει ως αρχή και πρόκειται την αρχή της αναλογικότητας. Ε, αυτό και εμείς το δανειστήκαμε και εμείς αυτό το επικαλούμαστε για τα όσο εμείς αποφασίζουμε. Θα το χρησιμοποιεί κάθε νομοθέτης, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι εάν θέλετε και εμείς να εφαρμόζουμε αρχή της αναλογικότητας, ε, τότε θα πρέπει να έχουμε την αναγκαία διακριτική, τραπέζη διακριτική ευχέρεια. Αυτό αφορά και για το MRL, αφορά τις σχετικές προθεσμίες ε, συμμόρφωσης και να δούμε το ότι δεν είναι ομοιογενής η κατάσταση σε όλες τις τράπεζες. Το θέμα είναι το κατά πόσον κάποια τράπεζα μπορεί να εξηγενθεί. Ε, τότε χρειάζεται το περιθώριο ε, ε, ελιγμόνο, ώστε το MRL να μπορεί να καλύψει την κάθε τέτοια περίπτωση. Οπότε βεβαίω και υπάρχει προσδοκία ε, ε, ε, αναλογικότητας, αλλά δεν μπορούμε ε, με, να υποχρεώσουμε κάποια, κάποια τράπεζα της φράσουμε Ζουρλομαδία το, το, το, μια κοινή μέθοδο. Επομένως, επομένως πρώτα πρώτα να μην θεωρούμε ότι ό,τι είναι σε μία υπόθεση και για τις άλλες και επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει διακριτική ευχέρεια ε, από πλευράς αρχής εξυγένσης. Τώρα όσον αφορά την ευελιξία για το πώς θα προσαρμοστεί, πού θα φτάσει το MRL και όσον αφορά τις αρχές εξυγίανσης θα πρέπει περιπτωσιολογικά να βρίσκουμε αν υπάρχει συμμόρφωση ή όχι τι γίνεται οπότε το σύστημα να γίνει κατά κάποιο τρόπο απλούστερο τώρα για το MRL επίσης πρέπει να κοιτάξουμε με φρέσκια ματιά τη λεγόμενη διαδικασία δύο επιπέδων. Οι στόχοι για το MRL καθορίζονται από το Συμβούλιο Εξυγέννηση. Εμεί απευθυνόμαστε σε εθνικέ αρχέ που πρέπει να εφαρμόσουν την απόφαση χωρίς να αφήσουν περιθώρια. Παίρνουν τη δική μας απόφαση και την εφαρμόζουν. Και αυτό σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο της καθεμιάς από τις 19 χώρες. Επομένως, θα πρέπει τελικά η απόφασή μας να έχει αποδέκεται στις τράπεζες. Έτσι θα ήταν πιο συμβατά τα αποτελέσματα ή η κατάρριξη αυτής της διαδρομής. Εδώ θα βάλω μια τελεία, ξέρετε εμείς τι χρειαζόμαστε για την φάση πριν την εξυγίαση η τόσο για την εξυγίανση με την ευρύτερη έννοια να μην μακρηγορώ και να καταλήξω κάπου. Όμως πρέπει να σας πω ότι το έντις την εγγύηση των καταθέσεων δεν θα την ε, θίξουμε η, το θέμα της ρευστότητα. Όμως δεν θα το θίξω τώρα. Αλλά στις ερωταπαντήσεις που θα ακολουθήσουν και το ίντις ε, θα το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ, λέει Σας ευχαριστώ για όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν με τις παρεμβάσεις. Πρώτος ο Μπορκάρτ Μπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε αυτό το μήνα την έκθεσή της για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και εκεί πέρα υπάρχει κάτι το οποίο είπατε το καλοκαίρι του 2016 και εκεί πέρα λέτε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί κάθε μήνα και χρόνο που περιμένουμε το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται είχατε κάνει αυτή την δήλωση πριν από δύο χρόνια ήδη και περιμένατε οπωσδήποτε πολύ εμείς Επίσης περιμέναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τώρα έχουμε τα σχέδια της Κομισιόν για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η έκθεση πρόοδου της Κομισιόν ε, επίσης ε, μιλάει για ένα επίπεδο 950 δισεκατομμυρίων ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα θέλαμε να δούμε και τα σχετικά νούμερα την ε, προηγούμενη εβδομάδα η Εποπτική Αρχή των Τραπεζών ε, μείωσε το επίπεδο φιλοδοξίας για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δατείων κατόπιν πολιτικής ε, πίεσης και μίλησε για μια ευκολότερη πρόσβαση στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με δημόσιο χρήμα, αλλά αν δεν ξεκαθαρίσουν τα πάλια χρέη και βάρη των ε, τραπεζών, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Γι' αυτό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σήμερα ποιες συμβουλές μπορείτε να μας δώσετε ως επικεφαλής ε, του Συμβουλίου Συντημικής Σταθερότητας για το ζήτημα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα μπορούσα εύκολα να πω πως ε, αυτό είναι θέμα των εποπτικών αρχών και όχι ε, δικό μου, αλλά δεν τα αποφεύγω. Είπα πολλές φορές και ισχύει αυτό όπως και στη συζήτηση για το Έμπρελ. Ε, για την ώρα η οικονομική κατάσταση είναι καλή, δηλαδή αν δεν δουν τώρα οι τράπεζες το ζήτημα ε, για να είμαστε ειλικρινεί, έχουν πέσει τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί ε, την πυθό τη, ε, κάποιοι λένε ότι λέει δύο κουβέντες εμπορικές, ε, ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Βεβαίως δεν θα βρεθεί μια λύση θαυματουργή και ανώδυνη. Οπότε το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε όντω το ζήτημα. Οι προτάσει τη Κομισιόν είναι πολύτιμε και περιλαμβάνουν ε, και ακριβώς ε, αυτό το οποίο είπαμε εμείς ε, για το τι θα γίνει ακριβώς με τις τράπεζες σε εθνικό υπερφυριακό επίπεδο αλλά δεν μπορούν να εξαφανιστούν με κάποιον μαγικό τρόπο οι ζημιές, ε, δηλαδή ότι αν υπάρξει κάποια κρατική χρηματοδότηση και κάποιο κρατικό όχημα θα εξαφανιστούν αυτά. Δεν εξαφανίζονται ως ε, διαμαγείας, ε, θα πρέπει ακριβώς να ξεχαρίσει το ζήτημα για την κάθε τράπεζα και νομίζω ότι Εντάξει, μπορεί η ΕΚΤ να πει ότι είναι λογικό να έχετε κάποια ιστορικά προβλήματα τα οποία πρέπει να εξαφανιστούν πριν περάσουμε στην επόμενη κρίση. Έχετε λοιπόν την στήριξή μας γιατί αν έρθει η επόμενη κρίση με αυτά τα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για να γίνει κάποια προληπτική διάταξη στην ε, νομοθεσία, αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι εξασθενούμε τις ε, διατάξεις, θα γίνει σωστά στην νομοθετική διαδικασία. Λοιπόν, Γιάκομπ Φων Βάιστσακε. Ευχαριστώ και κύριε Κένικ, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Ήθελα στην πρώτη με ερώτηση να επανέλθω στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου Νομίζω ότι μιας και βρισκόμαστε στη μέση της συζήτησης για τα MRL, χρήσιμο θα ήταν να έχουμε σχέδια εξυγίανσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων για να ξεκινήσουμε και να σταθμίσουμε καλύτερα την ε, μελλοντική μας αντίδραση, να δούμε και τι επιχειρήματα μπορούμε να προβάλλουμε για τα MRL και σε ένα ε, τοπίο που δεν επηρεάζεται μόνο πια από τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης. Άρα και δυστυχώς δεν ε, επηρεάζεται πια από το στόχο να βεβαιωθούμε ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι ε, χρηματοπιστωτικοί όμιλοι πρέπει να είναι σε θέση να διασωθούν, να εξηγιανθούν. Πώς λοιπόν μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι για τις πολύ μεγάλες τράπεζες θα προχωρήσουμε κάπως πιο γρήγορα Πώς μπορούν να έχουν πλήρως συμβατά ε, σχέδια εξυγένσης και τι διαδικασία μπορούμε να προβλέψουμε για την αποτίμηση, την αξιολόγηση. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει ο δικό σας οργανισμός ή κάποιος άλλος. Εάν τα πλήρως συμμορφούμενα αυτά σχέδια εξυγένσης ε, μπορούν στην πράξη να κάνουν ένα ίδρυμα απολύτως ε, δυνατό να διασωθεί, να εξυγενθεί. Δεύτερη ερώτηση για την αναθεώρηση και την ε, ερώτηση κατά πόσον θεωρείτε ότι μπορεί να το διαχειριστείτε και σε σχέση με όσα σας έχει δώσει η πείρα σας, να υπάρχει μια ε, μία μόνο αρχή εξυγένσης για τις μεγάλες περιπτώσεις. Ναι, για τις ερωτήσεις σας πρώτον, δεν έχουμε πλήρη συμμόρφωση ούτε πλήρη σχέδια εξυγένσης για όλες τις τράπεζες. Αυτό ισχύει για δύο λόγους και εν μέρη γιατί οι μεγαλύτερες τράπεζες ήδη έχουν ένα σημαντικό επίπεδο MRL. Όταν λοιπόν λέμε ότι θέτουμε στόχους για τα MRL, χοντρικά οι μισέ από τις τράπεζες που δεσμεύονται από στόχου για MRL του ακολουθούν. Μπορεί να αυξηθούν οι στόχοι που του θέτουμε με τον χρόνο, αλλά περίπου οι μισέ δεν χρειάζονται καμία περίοδο μετάβασης. Διότι ήδη ε, το μέρος του, ένα μέρος του στόχου του το έχουν πετύχει Βεβαίω είναι πύριο νίκη γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά κάποιε τράπεζε είναι ήδη σε καλή θέση. Μερικές άλλες χρειάζονται περίπου δύο χρόνια στο, πρόγραμμα, στο σχέδιο προγραμματισμού τους για να προχωρήσουν. Για άλλες θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και για κάποιες άλλες είναι πιεστικά τα πράγματα. Μπορεί να προκύψει αυτό. Εάν δεν έχουμε την απαιτούμενη ποιότητα MRL, η δυνατότητα εξυγίανσης δεν θα είναι κάτι το προφανές για τις τράπεζες αυτές. Είναι ένα ταξίδι που θα συνεχιστεί. Για το κατά πόσο το πρόγραμμα εξηγήσεις κάνει την τράπεζα πραγματικά σε να, να είναι σε θέση να εξηγιανθεί, το σώμα των ε, υπευθύνων των φορέων θα αποφασίσει σχετικά. Δηλαδή υπάρχουν και υπεύθυνοι για τη διάσωση και την εξυγέννηση εκτός Ευρωζώνης και τελικά αυτοί λαμβάνουν την απόφαση. Πάντως τους στόχους του θέσαμε το 2017 ήταν μια πρώτη φάση της πορείας αυτής και θα πρέπει να υπάρξουν και περισσότερες. Ε, περισσότερο στην, στην άποψη της ποιότητας και μετά και της ποσότητας για την αναθεώρηση ευθύς εξ αρχής έχω την αίσθηση ότι για τις μεγάλες για τις μεγάλες ε, τράπεζες, στις, στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, περισσότερες έχουν ήδη διεθνή δράση για να τις έχουμε στον τομέα της ε, κατάστασης και εξυγένσης είναι λίγο δύσκολο. Για μένα θα ήταν πολύ λογικό, αλλά δεν το αποφασίζουμε εμείς. Είναι ένα πρώτο βήμα να μιλήσουμε πρώτα για την ανάκτηση και μετά για την εξυγίανση. κεντρική αντισυμβαλόμενη. Όμως είναι μέρος του οικοσυστήματος των τραπεζών και δεν μπορούμε να, τις, ε, να αντιμετωπίσουμε ανεξαρτήτως. Εκτιμούμε λοιπόν τη ρήτρα αναθεώρησης και θα πρέπει να το κοιτάξουμε περαιτέρω. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λούκε, όχι, ο κύριος Ζήλε. Ναι, ναι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ο Ραμόν Τρεμόζα. Ο Ραμόν Τρεμόζα καλώς ήρθατε και πάλι. Ε, έχω κάποιες ερωτήσεις. πρώτη αφορά τις Ιταλικές εκλογές. Ανησυχείτε για το ότι κέρδισε τις εκλογές ένα κόμμα που είναι κατά του Μπεϊλίν. Έχετε κάποιο σχόλιο. Δεύτερη ερώτηση για την ε, λετωνική τράπεζα, η BLB. Την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΚΤ έκρινε ότι η τράπεζα αυτή και η θηγατρική της στο Λουξεμβούργο θα χρεοκοπούσε. Όμως ε, αποφάσισε το Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας ότι δεν ήταν προς το δημόσιο συμφέρον μια διάσωση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε να μου πείτε γιατί. Τρίτον, ποια είναι η επίπτωση της απόφασης του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου για την λύση της ε, θύγατρη, το κλείσμα της θηγατρικής εταιρεία αυτής ε, στο Λουξεμβούργο και την προηγούμενη φορά μας είπατε, ε, είπατε στην Ισπανική Εξεταστική Επιτροπή πως η τελική αξιολόγηση της Deloitte για την Banco Popular θα ήταν διαθέσιμα οι αρχές του 2018. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα δημοσιευτεί. Γιατί ξέρετε ότι ο σχετικός κανονισμός λέει ότι το Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας λέει ότι θα πρέπει αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Και ήταν αυτό πριν από εννέα μήνες. Να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Είπα στην εισαγωγή μου πως εμείς όπως και εσείς περιμέναμε την αξιολόγηση αυτή. Περίμενα να υπάρχει τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο. Δεν έχει τελειώσει ο Μάρτιος, αλλά πρέπει να είμαι επιφυλακτική. Η αξιολόγηση είναι ανεξάρτητη και είπαμε ότι θέλουμε να υπάρξει αυτή η εκτίμηση ακριβώς ε, το συντομότερο δυνατόν, αλλά δεν την συντάσσουμε εμείς και δεν ε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να του ζητάμε τώρα. Έχω ακούσει Απρίλιο, αλλά πρέπει να είμαι επιφυλακτική, γιατί πριν μου είχαν πει Φεβρουάριο. Το δεύτερο θέμα, Ιταλικές εκλογές. Όπως και εσείς ε, παρακολουθώ τις εκλογές στα κράτη-μέλη και οι ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται. Τώρα θα σχηματιστεί η κυβέρνηση και θα δούμε. Δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο για την τράπεζα της συγκεκριμένη Λετωνίας, για να είμαι σαφής. Μαζί με τους συναδέλφους μας ε, στο εθνικό επίπεδο, από τη Λετωνία δηλαδή, και από το Λουξεμβούργο, ήδη το 2017, το 2016 μάλιστα, είχαμε συζητήσει και λέγαμε ότι η τράπεζα δεν, είναι, δεν έχει συστημική σημασία για την λετωνική οικονομία ούτε για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν απειλεί την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. Ο λόγος ε, είναι πως ε, είχε ένα περίεργο επιχειρηματικό μοντέλο. 80% των καταθέσεων της τράπεζας ήταν καταθέσεις από ε, πολίτες τρίτων χωρών. Κατά κύριο λόγο Ρώσους, Ουκρανούς από την κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών, εν πάση περιπτώσει. Και άρα είχε και μικρή συνδεσιμότητα εντός της οικονομίας της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς ε, καταλήξαμε όταν ελήφθη αυτή η απόφαση ότι ε, συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σχέδιο εξυγίανσης. Και μετά είπαμε πως ε, θα έπρεπε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εξυγίανσης, αλλά βεβαίως οι κατατόπους νόμοι είναι εθνικοί και μια που έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, το δικαστή, τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου αποφάσισαν βασιζόμενοι στο ότι η τράπεζα είναι φερέγγια, έχει επαρκή κεφαλαιοποίηση, είναι και πολύ μικρή η τράπεζα έχει καλά στοιχεία ενεργητικού, απλά δεν έχει ρευστότητα γιατί δεν, δεν μπορεί να ρευστοποιήσει τα στοιχεία που έχει σε δολάρια. Γι' αυτό τους επιτρέπει ένα χρεοστάσιο, αλλά δεν θεωρεί ότι είναι σε θέση να ε, κηρύξει την τράπεζα υποπτώχευση. Αυτή είναι μια απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Στη Λετωνία η κατάσταση είναι διαφορετική. Εκεί ε, η τράπεζα πήγε, η διοίκηση δηλαδή, εθελοντικά σε μια διαδικασία χρεοκοπίας ε, η οποία αυτή τη στιγμή αξιολογείται και μάλλον θα περάσει, θα εγκριθεί. Οπότε το δίδαγμα είναι η εναρμόνιση αυτού του τμήματος του πτωχευτικού δικαίου θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζήλε, θέλετε τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς ε, αυτό ήταν το ε, τμήμα μιας ερώτησής μου, αλλά ε, δυστυχώς συνεδριάζουν δύο επιτροπές παράλληλα και πρέπει να είμαι σε δύο μέρη. Σας ευχαριστώ. άκουσα τμήμα της απάντησής σας, είμαι από τη Λετωνία, ήθελα και εγώ λοιπόν να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα με την τράπεζα αυτή, την ABLB, αλλά Έχω και ένα παρόμοιο θέμα. Η τράπεζα αυτή είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια πολιτική απόφαση, οπότε δεν, ότι δεν έχει συστημική σημασία. Στην ε, περίπτωση αυτήν ε, δεν υπήρχε δημόσιο συμφέρον στο να συνεχίσει να λειτουργεί η τράπεζα. Γι' αυτό ακριβώς ε, δεν ενεργοποιήθηκε ο σχετικός μηχανισμός. Μπορούμε σε αυτήν την περίπτωση βλέπουμε ότι και η πρώτη και η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα σε ένα μικρό κρατός μέλος Ευρωζώνης ε, δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα συστημικό στην Ευρωζώνη. Συμφωνείτε και αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που προκύπτει εδώ πέρα ειδικά στην περίπτωση όπου τα πράγματα είναι στα χέρια κρατών μελών ε, όπου ο τραπεζικός τομέας ε, έχει μεγάλη σχέση με κατοίκους τρίτων χωρών και έχει μεγάλη σημασία το θέμα του ξεπλήματος ε, χρήματος και όλα αυτά φαίνονται αυτομάτως στον ισολογισμό της τράπεζας. Θεωρείτε ότι πρέπει λοιπόν ε, η καταπολέμηση του ξεκρεπλήματος χρήματος να αφαιρεθεί από τα κράτη-μέλη και να πάει στην ΕΚΤ τουλάχιστον για τις μεγαλύτερες τράπεζες ε, της αγοράς. Η ερώτησή σας σημαίνει ότι η πρώτη ή η δεύτερη τράπεζα σε ένα μικρό κράτος μέλος δεν θα ε, μπορούσε ποτέ να φτάσει σε κατάσταση να εξηγενθεί. Όχι. Θα έλεγα ότι έχουμε ένα σαφές όχι ως απάντηση. Η ABLB ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ήταν αυτό το οποίο εξήγησα. 80% των καταθέσεων αφορούσε ε, ανθρώπους που δεν ήταν κάτοικοι της ε, χώρας. Οπότε μπορούσε να πει κανείς πως δεν είχε μεγάλη ε, σχέση με την οικονομία της χώρας, ούτε με τα νοικοκυριά, ούτε δάνεια σε επιχειρήσεις της χώρας. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι επειδή ε, με βάση τα ευρωπαϊκά μεγέθη είναι μικρή τράπεζα ότι αυτό ήταν ο λόγος. Και αυτή ήταν μια απόφαση την οποία λάβαμε σε απόλυτη συμφωνία με τους συναδέλφους της Λετωνίας ε, και του Λουξεμβούργου. Η επόμενη ερώτηση τώρα για να περάσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα ξεπλήματος χρήματος δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν το κάνουμε εμείς ούτως ή άλλως. Σαφώς υπάρχουν υπέρ και κατά και αν δει κανείς την κατάσταση υπάρχει το μεγάλο συν ότι οι υποπτικές αρχές έχουν και μεγαλύτερο λόγω όσον αφορά ακριβώς τον κίνδυνο της φήμης σε σχέση με το τι έχει σήμερα. Σας ευχαριστώ, Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Άρα έχουν περάσει περισσότερα από τρία, τα τρία χρόνια που δημιουργήθηκε το Συμβούλιο και οι υπόλοιποι φορείς της Τραπεζικής Ένωσης. Και πολλοί ρωτούν το εξή. Στην Ιταλία δεν ότι τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Πάλι δόθηκε κρατική βοήθεια. Ενώ είχαμε πει ότι θα πάυσουν οι επιδοτήσεις της Τράπεζας της Ένωσης. Είχαμε την υπόθεση Banco Popular που μάθαμε ότι τα στοιχεία που είχε το Ίδρυμα στα χέρια του για να αντιμετωπίσει το θέμα ήταν τελείως ανεπαρκή. Και είσαστε και τυχεροί που βρέθηκε κάποιος για να πληρώσει για το θέμα και τελικά σωθήκαμε. Τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και άλλο πρόβλημα γιατί μια σχετικά μικρή τράπεζα στην Λετωνία ε, πάει για πτώχευση λόγω θεμάτων ξεπλήματος χρήματος. Οι αρχές δεν συμφωνούσαν εάν θα αποκαλέσουν την τράπεζα τράπεζα σε πτώχευση ή πιθανόν απτωχεύση. FOLTF. Τελικά πότε λειτουργεί το σύστημα, πότε είναι τα πράγματα φυσιολογικά και ισορροπημένα και πάνε όλα καλά όπως υποσχεθήκαμε στους πολίτες και τι μπορείτε να μας πείτε σε εμά ως ε, συνομοθέτες ώστε το σύστημα τελικά να λειτουργήσει. Θα ήθελα να μου πείτε ένα κατάλογο από τις επιθυμίες σας, τις υποτεραιότητές σας και τον καλωσόριζα. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Απλώς να διευκρινίσω το εξής, ότι στην περίπτωση της Banco Popular δήλωσα κάποια στιγμή ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση συνειδητοποιήσαμε ότι τα δεδομένα, τα στοιχεία θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά δεν δημιούργησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το θέμα αυτό λύθηκε η Banco Popular μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά, ως παράδειγμα για πολλά θέματα, για πολλές περιπτώσεις, αλλά βάσει του ε, βιβλίου κανόνων βρέθηκε ε, αγοραστής. Ε, αν δεν είχε βρεθεί θα υπήρχε θέμα χρηματοδότησης, κάλυψης της, ανάγκης να διασωθεί τώρα για τη Λετωνική Τράπεζα και τον κατάλογο με τις επιθυμίες μας, ε, αυτό που ε, ισχύει είναι ότι υπάρχει το σύστημα διάσωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και εξυγίανση, αλλά υπάρχει και το θέμα τη πτώχευση που ρυθμίζεται σε εθνική, στην εθνική νομοθεσία. Άρα, εδώ έχουμε μια τράπεζα που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έχουμε μια απόφαση για σεπτόχευση ή πιθανόν απτοχεύση, αλλά δεν είναι εύκολο η απόφαση αυτή για FOLTF να μεταφραστεί εύκολα σε εθνική νομοθεσία και να συνδυαστεί με του σχετικού κανόνε πτώχευσης. Για τον κατάλογο με επιθυμίας μας αυτό που θέλουμε να γίνει είναι να κινηθούμε με ταχύτητα και να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι κατάλογος επιθυμιών, είναι κατάλογο ε, προ εκπλήρωση υποχρεώσεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευελιξία αλλά και ρεαλισμό. Δηλαδή να ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσουν όλα να γίνουν ε, στην εντέλεια μέσα σε ένα χρόνο. Χρειάζεται χρόνος. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να κινηθούμε στη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσα να σας ε, παρεθμίσω έναν μακροσκελή κατάλογο επιθυμιών όμως ήδη τα θέματα της χρηματοδότησης, της οικονομικής κάλυψης και της εξυγίανσης είναι ένα θέμα. Μετά θα μπορούσαμε να έχουμε και την brd 2 σε λειτουργία. Είναι ένα νομοθετικό πακέτο που μπορεί να αλλάξει τελείως το όλο τοπίο και αυτό είναι μέρος των επιθυμιών μας. Νομίζω ο γιος μου είναι πολύ πιο ανοιχτό ό,τι αφορά τον κατάλογο των επιθυμιών του και πολύ πιο απαιτητικό. Σα παρακαλώ να είστε και απαιτητικοί μαζί μα. Θα είμαι. Είσαστε πολύ απαιτητικό εσεί. Αυτό είναι ο ρόλο μου εδώ σε αυτή την επιτροπή. Τι να κάνουμε, πρέπει να εφαρμόσουμε το ένα ή το άλλο από την νομοθεσία. Έχουμε συζητήσει διαμακρών για το θέμα αυτό, δεν θα συνεχίσουμε τώρα. Ο κύριος Σίντερεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κένικ που ήρθατε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Για μια μικρή πολιτική ομάδα όπως η Γκουε είναι συχνά δύσκολο να επιβληθεί στο Κοινοβούλιο, αλλά Βεβαίω οι αρμοδιότητές σας ε, ε, βρίσκονται νομίζω αρκετά κοντά στις δικές μας επιθυμίες. Έχουμε και εμείς κάποιες επιθυμίες. Λοιπόν, οι δικές μου ερωτήσεις έχοντας ακούσει και τους ε, συναδέλφους ελπίζω να σας δώσουν την ευκαιρία να επεκταθείτε. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά σε αυτό το οποίο αναφέρατε για την επεξεργασία της οδηγίας BRRD. Ένα θέμα συζήτησης μεταξύ των πολιτικών ομάδων είναι ακριβώς το πώς θα οριστεί αυτό το περιθώριο MRL για την κάθε τράπεζα και το θέμα είναι αν θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ευστηρότεροι κανόνες. Και κατά την άποψή σας η πρόταση της Κομισιόν πηγαίνει στην σωστή κατεύθυνση ή θέλετε περισσότερη ευελιξία για το Συμβουλίο σας για να υπάρξει επαρκής διασφάλιση. Μια δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω σχετίζεται με το εάν θεωρείτε πως θα πρέπει τα MRL να βρίσκονται ε, υποτεταγμένα σε σχέση με άλλα χρήση. ευχαριστώ σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ε, να συμφωνήσω. Για την ε, PRD2 ε, και το αρχικό πακέτο, δύο, δύο ήταν τα θέματα που είχαν σχέση με τα MIL. Πρώτα απ' όλα οι αυστηρές απαιτήσεις... για G-SIPs και άλλες για O-SIPs και τις άλλες σημαντικές συστημικές τράπεζες. Ήταν οι ελάχιστες απαιτήσει για τα επιμέρους κράτη-μέλη των G-SIPs, κάτι που μας απασχολούσε πολύ και μετά η κρίση δεν είναι τα MRL μαθηματικός υπολογισμός από μόνα τους. Ο στόχος είναι να, είναι σε να, να είμαστε σε θέση να διασώσουμε τις τράπεζες με αυτά. Γι' αυτό πρέπει να τοποθετηθούν στην πολύπλοκη οργάνωση ενός ομίλου, να ε, ληφθούν υπόψη στο, στην όλη δομή του ομίλου και μας ενδιαφέρει να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας τα MRL, γιατί ε, επιλύουν το πρόβλημα του κανένας πιστωτής δεν βρίσκεται σε χειρότερη θέση, no creditor worst off, διότι οι senior ε, πιστωτές δεν καλύπτονται ούτε διασώζονται ε, εάν πρόκειται να δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα χωρίς να δημιουργούμε ένα άλλο. άρα, για να χρησιμοποιήσω και την έκθεση του κ. Ε, είναι ένα κατάλογο επιθυμιών αυτό, αλλά χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και ακόμη περισσότερο σαφήνεια. Σαφήνεια για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εσωτερικών, Εμαριέλ, μέσα σε έναν όμιλο. Μπορεί δηλαδή να μιλά κανεί για Μαριέλ σε έναν όμιλο, αλλά εσωτερικό πρέπει να τα τοποθετήσει σωστά. Δηλαδή μερικά πρέπει να μπουν στη σωστή θέση, μερικά άλλα πρέπει να προτοποθετηθούν. Είναι πολύ δύσκολο γιατί γίνεται τμήμα ανά τμήμα και πρέπει να μην είμαστε και υπέρμετρα φιλόδοξοι ανάλογα με τις διαστάσεις του κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και ομίλου. Ευχαριστούμε ο κύριος Βάλλη νίκησε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Ραμόν. Μη φοβάστε τόσο πολύ τη λαϊκή ψήφο. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα σε σχέση με τη σύγκρουση σφαιρόντων των λεγόμενων ανεξάρτητων αρχών. Εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια. Δύο ερωτήσει προ εσά, κυρία Κένινγκ. Πρώτον, προσπαθείτε να λάβετε υπόψη στις ε, εκτιμήσει που θα γίνουν για τα MRL τα διάφορα μοντέλα υπολογισμού του πιστοτικού κινδύνου που υπάρχουν εντός του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε σε τι πλαίσιο κινείστε και με τι περιθώριο διακριτικής ευχέρειας. Και μετά, τι ε, εμπειρίες έχετε αποκομίσει σε σχέση με τη ρευστότητα τα MIL είναι ένα πρόβλημα, αλλά εδώ έχω κάποια στοιχεία που μας ανησυχούν. Έχουμε τα 950 δις ευρώ αγορά του, στην αγορά των ε, MRL, παραγόγων ε, ή τέλο πάντων MRL, ε, μιας αγοράς που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανωδική πορεία, αλλά μπορεί να εξαντληθούν ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε λοιπόν 6.700 ε, εκατομμύρια και 453 όπου πρέπει να Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ε, σκεφτούμε την σύγκρουση συμφερόντων σε αυτήν την κατάσταση που μπορεί να είναι προβληματική όμως ε, εδώ να είμαστε και βέβαια ότι δεν ξεχνάμε κανένα τομέα εκτός. I not... Σας διαβεβαιώνω ότι δεν τα ξεχνούμε. Αλλά ξέρετε, στο παρελθόν τα έχουμε ξανασυζητήσει. Πρώτα απ' είναι θέμα του εποπτεύοντος να αξιολογήσει τον ε, κίνδυνο για τις πιστώσεις και σε σχέση με τις κυβερνητικές απαιτήσεις. Εμείς ασχολούμαστε και με τα παραγόγα, με τη ρευστότητα του ενεργητικού, ε, για την δυνατότητα για περιθώρια εξυγίανσης. Προσπαθούμε όλα αυτά να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και συμμετέχουμε εμείς και άλλοι σε αυτή την προβληματική για να δούμε τελικά τι θα γίνουν, πώς θα έχουν αίσια εκαθάρισε κάποια χαρτοφυλάκια παραγόγων. Ναι, όλα αυτά είναι στο έργο μας, αλλά θα πρέπει να δούμε από πλευράς αξιολόγησης τι κάνει ο αξιολογητρικό. Νομίζω ότι καλά τα πάει. Και να δούμε τι θα αξιολογήσουμε εμείς όταν έρθει η ώρα να κάνουμε την ούτως κατάτμηση. κατάτμιση σε χαρτοφυλάκια κάποια τράπεζα στην περίπτωση τη εξυγίανση. Thank you. Um, Barbara Η κυρία Καπέλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύρια Κένικ ε, και για αυτά τα οποία είπατε για το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων και το MPL και είπατε σε μια συνέντευξη τον Φεβρουάριο πως θέλετε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων παρά το ότι είναι επίμαχο θέμα σε κάποια κράτη-μέλη, ειδικά οι εκπρόσωποι των γερμανικών ταμιευτηρίων και συνεταιριστικών τραπεζών ζητάνε να υπάρξει μείωση των κινδύνων πριν περάσουμε σε ένα διαμοιρασμό των κινδύνων. Ταυτόχρονα είπατε πως είστε κατά του bailout και η Κομισιόν είπε πως θα υπάρξει ένα σχέδιο δράσης για την μείωση ακριβώς ε, των κινδύνων αυτών ε, και ακριβώς ε, το πώς θα υπάρξει και μια αλλαγή είτε του κανονισμού περί ιδίων κεφαλαίων είτε κάτι θα πρέπει να γίνει δευτερογενείς αγορές. Ε, και μιλήσατε επίσης στην τελευταία έκθεση προόδου για μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τάξης των 900 δισεκατομμυρίων, μη εξυπηρετούμενα της τάξης των 900 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εάν λοιπόν υπάρξει μια κοινή εγγύηση των καταθέσεων πριν ε, υπάρξει μία μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τίθεται ένα ερώτημα. Κάποια κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Ιταλία, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν λάβει καθόλου επιπλέον μέτρα για να μειώσουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μήπως λοιπόν έτσι θα αυξηθεί ο συστημικός κίνδυνος για τις ε, τράπεζες αυτές. Σας ευχαριστώ να προσπαθήσω να απαντήσω την ερώτηση και να εξηγήσω γιατί προτείνουμε όχι σήμερα ε, άμεσα ένας ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης κατανθήσεων. Αν δείτε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχουμε έναν ενιαίο μηχανισμό αναδιάρθρωσης και εποπτικό μηχανισμό. Και με ρωτήσετε για το MREL. Και στο MREL πάντα συζητάμε τι, πώς γίνεται και τι θα γίνει από την πλευρά της χώρας υποδοχής εάν χρεοκοπήσει μία τράπεζα και κάποιος ξεχάσει την θηγατρική της σε άλλη χώρα. Τότε υπάρχει ένα εθνικό πρόβλημα και αν πάντα πράγματα στραβά η καταθέσεις ε, θα είναι εγγυημένε σε εθνικό επίπεδο. Οπότε το δικό μα το επιχείρημα είναι, αν θέλετε πραγματικά να έχουμε μια τραπεζική ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα πρέπει και το σύστημα εγγύησης ε, των καταθέσεων ή το σύστημα εξυγένσης να είναι ευρωπαϊκό για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν λανθασμένα κίνητρα ή κάποια εθνική ε, προκατάληψη. Τώρα συμφωνώ ότι αφενός θα πρέπει ε, μαζί με τη μείωση κινδύνου να πάει χέρι-χέρι να πάει χέρι-χέρι μείωση κινδύνου με τον από κοινού διαμοιρασμό του κινδύνου, αλλά δεν συμφωνώ στο ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το έχουν δει τα κράτη-μέλη, μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να λέμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και πιο γρήγορα. Και έτσι θα έλεγα ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία έχει κάνει η Κομισιόν και η ΕΚΤ τους τελευταίους 12 μήνες. Έχουν αυξήσει την πίεση και λένε πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το θέμα. Θα δούμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι θα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί κάτι και να περάσουμε στην επόμενη φάση ή προσπαθούμε να κινηθούμε κάπως ε, και νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν ήταν τουλάχιστον ένα βήμα. Ας δούμε πώς θα πάει η συζήτηση, αλλά τελικά το σύστημα χρειάζεται και τα δύο σκέλη. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Ντανούτα Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως πάντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας ακούμε κύριε Κιονίκη. θέλω να ξαναγυρίσουμε στο Τίλεκ e και στο MRL. Αλλά να δούμε τι θα γίνει μετά από τον Brexit. Τότε όλα αυτά τα εργαλεία και μέσα του Βρετανικού Δικαίου πλέον δεν θα καλύπτονται από το ΤΙΛΑ και το MRL. Δεν θα υπάρχει συμβατική ρήτρα που απαιτείται από το 55. Οπότε σας ερωτώ, τι λύση θα δοθεί για τις νέες συμβάσεις αλλά και για όσον ακόμα εκκρεμεί η λύση. Επίσης, για πέστε μας για αυτό το μνημόνιο που λοιπόν, αναφέρατε για το με του BRRD. Τι είπατε? Ο μορατόριο, μορατόριο όμως. Α, ναι, το μορατόριο όμως είναι πιο ωραίος λέξη. Λέει η κυρία Χούμπνα. Και για αυτό το χρεωστάσιο. Πολλές πολιτικές ομάδες εδώ έχουν ασχοληθεί σε σχέση με την διάρκεια αλλά και για το ότι ίσως αυτό το μέσο δεν είναι το πιο δόκιμο αλλά ακούμε όμως ότι ο πλευράς ε, αξιολογητή είναι. Εσείς πώς το βλέπετε. Σας ευχαριστώ. Για να σας πω πρώτα πρώτα για το Brexit. Πέρσι αρχίσαμε και το συνεχίζουμε φέτος να λέμε στις τράπεζες ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για τα χειρότερα. Για τα χειρότερα θα ήταν ότι μετά το Brexit ό,τι ίσχυε δυνάμει του λόγου του Ηνωμένου Βασίλου, του Βρετανικού Δικαίου, τώρα δεν θα καλύπτεται από το MRL. Έχουμε ασοροσυμβετικές ρήτρες, αλλά ό,τι εκδοθεί τώρα θα έχει μία σχετική ρήτρα. Εγώ θα προνούσα να υπάρχει νομοθετική αναγνώριση όπως τώρα ε, ισχύει στην ε, Βρετανία. και υπάρχει αμοιβή αναγνώριση, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε προ το παρόν είναι να πούμε ότι το ελάχιστο που απαιτείται να υπάρχει μια συμβατική ρήτρα γιατί πια δεν θα υπάρχει νομοθετική κάλυψη και ότι η νομοθετική κάλυψη υπήρχε πριν θα αντικατασταθεί από άλλη. Τώρα όσον αφορά αυτό το δεύτερο χρεοστάσιο Εμεί θεωρούμε ότι ισχύει το δεύτερο εργοστάσιο, όχι πάντοτε, αλλά στην εργαλειοθήκη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και ίσχυσε για την Λετωνική Τράπεζα, ούτω ώστε η τράπεζα να μπορεί να έχει την αναγκαία ρευστότητα ή να την δημιουργήσει και να μην κλείσει η τράπεζα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις και εμείς ως αρχή διάσωσης εξηγήνωσης θεωρούμε ότι για αυτές τις ε, αποφάσεις failing like to fail να δώσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια ευκαιρία και σε σχέση με την απόφαση της διάσωσης του ώστε να μπορεί να μείνει η τραπέζα το Σαββατοκύριακο. Να είναι ευρεία η χρήση του ή το να καλύψει και τις καταθέσεις, δεν θα μπορέσουμε να φρενάρουμε την εκροή του χρήματος. Καλά είναι πέντε μέρες μεταξύ του ενός και του άλλου, αλλά τέλος πάντων, εγώ πάντα λέω ότι θα πρέπει να το εφαρμόζουμε με την ευρία έννοια. Και οι τράπεζες ακριβώς έχουν αυτές τις αλήτρες ε, και τα πρωτόκολλα. Όλα αυτά σε κάποιο δεύτερο χρηστάσιο θα μπορούσαν να καλύπτονται ως παρεκκλήσεως εξαιρέσεις. Αλλά για να το πω, μα αυτό είναι ένα εργαλείο χρήσιμο σε περιπτώσεις μικρού ελληνικού. Εντάξει, Ντανιέλα, δεν με εξέλιξε παντός η ερώτησή σου. στους Μπερές. Ευχαριστώ. Για να επανέλθουμε στην υπόθεση της ε, Λετονικής ε, Τράπεζας. Και γιατί ακόμα δεν διαπιστώσαμε, δεν συνειδητοποίησαμε τι έγινε ε, με τον SSM. Γιατί γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Και για την Ιταλική και για την Ισπανική υπόθεση. Υπήρχαν ερωτηματικά σε σχέση με το πώς μεταδόθηκαν κάποιες πληροφορίες μεταξύ SSM και SRB. Τώρα όμως ε, θα πρέπει να δούμε τι συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και είπατε ότι θα πρέπει να εξετάσετε το θέμα της φήμης της τράπεζας ότι και αυτό θέλετε να το εξετάσετε. Έτσι απαντήσατε προηγουμένως σε συνάδελφο. Στον κανονισμό χρησιμοποιείται μία φορά η λέξη φήμη. Αλλά όχι όπως το χρησιμοποιήσατε εσείς. Άρα, τι θα κάνετε στο μέτωπο αυτό. Πώς θα παρακάμψετε το αδιέξοδο στο οποίο έχετε βρεθεί. Αν λέτε ότι θα πρέπει να υποπτεύσετε, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική των ε, τραπεζών σε σχέση με το ξέβλημα χρήματο, μια που δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά θα πρέπει κάπως να βρείτε τρόπο παράκαμψης για να μπορέσετε να το καλύψετε. Να, επικαλείστε το, την έννοια της ε, φήμης, business model έχετε πει άλλη φορά αλλά τι συγκεκριμένα θα κάνετε. Και για τις επαφές με το SSM ε, και σχέση με το SSM τέλο πάντων και αυτό είναι κομμάτι της εργαλειοθήκης. Χρειάζονται καθεντήριες, χρειάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας. Άρα τι ίσχυσε εσύ για τις πληροφορίες ε, που έχουν σχέση με την Λετωνική Τράπεζα. Γιατί πρόκειται τώρα για, για θέμα κατανομής αρμοδιοτήτων κρατών και ένωσης. Για την πρώτη σας ερώτηση για τη σχέση μεταξύ SSM και SRB στην υπόθεση της Λετωνικής ε, Τράπεζας, όπως είπαμε, βασικά ενημερωθήκαμε ταυτόχρονα με, τα, με, με, με, με την ανακοίνωση τύπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγε ότι είναι ιδιαίτερος ε, η υποπτή αλλά ότι ακόμα η τιμιγορία ούτως υπήν δεν έχει διαμορφωθεί τώρα σε σχέση με τον SSM είχαμε πολύ στενή συνεργασία άρεστη συνεργασία αυτή εξ αρχής για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα επομένως με τίποτα δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε πρόβλημα. Και όπως έλεγα επίσης, δεν αποτελεί κριτήριό μας η φήμη για το να δούμε κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος που έχει Είναι θέμα περισσότερο του SSM και όχι δικό μας. Όμως πάντοτε λέω στο προσωπικό μας να μην συγκατανεύεται, να μην ε, μην αδιαφορείτε τέλος πάντων όταν βλέπετε καλά στοιχεία σε μια τράπεζα. Κοιτάξτε και πέρα από αυτά το business model, τι κάνει η τράπεζα ακριβώς. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Μιαν, ανοίξει και γρήγορα το κουτί της Πανδώρας με τις εκπλήξεις. Ε, φυσικά όμως και αυτό είναι θέμα SSM και όχι δικό μας. Εκεί, εκεί εμπίπτουν όλα αυτά τα θέματα, το business model, διαχείριση και αυτά. Εμεί περιζόμαστε στο πλάνο της εξυγίνησης της διάσωσης. Τώρα όσον αφορά με το θέμα του ξεπλήματος ε, προϊόντων εγκλήματος, αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Τα κράτη-μέλη κάνουν την επιλογή ή αν θα πασάρουν το θέμα δηλαδή στην Ευρώπη ή αν θα λύσουν το θέμα μόνο τους. Τώρα, το αν χρειάζονται κατευθυντήριες ή νομοθέτημα, εντάξει, ήταν κάπως ε, μαγνωμένη αυτή η περίπτωση. Απλώς περιπτωση απλώ επρεπε να ξυπνήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε κατά πόσον υπάρχει κάποια απειλή την τράπεζα, να χτυπήσουν το, με τον συναγερμό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος I... Ευχαριστώ ε, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στη χώρα μας. Πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ξεπεράσαμε την ε, κρίση του 2015, αργά αλλά σταθερά, αλλά ακόμη παραμένουν προβλήματα. τα MRL είναι σε χαμηλό επίπεδο, το ίδιο και κατεθέσει. Πώ αντιμετωπίζετε λοιπόν η κατάσταση, υπάρχει ένα σύστημα εγκύρης προειδοποίηση. παρακολουθείτε το πώ εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες, υπάρχουν ειδικέ διατάξεις, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Πάντοτε προσπαθώ να μην σχολιάζω ε, ξεχωριστά τις διάφορες χώρες αλλά αν δείτε τις αποφάσεις μας για τα MRL και τα προγράμματα διάσωσης και εξυγίανσης του 2017 στην στατική μας δηλώναμε ότι δεν θα λάβουμε δεσμευτικές αποφάσεις για τράπεζες που ακόμη βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης για τις οποίες η επίτευξη των MRL δεν είναι κάτι το επικείμενο. Δεν επίκειται. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάθε τράπεζα που θα μπορούσε να πτωχεύσει και να χρειαστεί εξυγένση χρειάζεται η ΑΕΛ ούτως ή άλλως. Είναι λοιπόν μια πορεία σταθερή. Αυτά μόνο μπορώ να πω. Ευχαριστούμε ο κύριος Φερνάντες. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, bienvenida al... Σας ευχαριστούμε και καλώς ορίσατε. Πρώτα πρώτα και εγώ να συμφωνήσω. Έχετε δίκιο να είσαστε ανυπόμονοι. Όπως και όλοι οι συνάδελφοι που είναι ανυπόμονοι όσον αφορά την ε, έκθεση της ε, Deloitte, Deloitte τέλος πάντων, όσον αφορά την μεταχείριση του, των ε, οφειλετών. Ναι, εντάξει, ας ασκηθεί λίγο παραπάνω πίεση για να τα μάθουν ώρα Τώρα, τώρα, για την Λετωνική Τράπεζα, ABLV, σταθήκατε στο ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε, να εναρμονίσουμε τα πτωχευτικά δίκαια για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση του αν ε, πρέπει να εξηγενθεί και να καθαριστεί μια τράπεζα. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει κάποιο είδου κοινή ασφάλιση των καταθέσεων Όπω ξέρετε έχουμε 19 διαφορετικά καθεστώτα και σε μερικέ χώρες έχουμε και παραπάνω από ένα σύστημα για τι καταθέσει. Διαφορετικέ πολιτικές, διαφορετικά μέσα πολιτική. Ε, αυτό είναι ένα παραπάνω πρόβλημα όταν έρχεται η ώρα να αξιολογηθεί το ποια θα είναι η μοίρα προβληματικής τράπεζας. Πώς βλέπετε την πορεία των ερμαντεύσεων για το σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων. Πώς βλέπετε κάποιες προτάσεις που αφορούν την ε, αντασφάλιση κάποιων εθνικών ε, ασφαλίσεων. Γιατί από το 2014 και μετά έχουμε μια συναλλαγή για τα χρέη που είναι από τράπεζα προς τράπεζα και δεν υπάρχει κάποιο είδους ισότιμη βάση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο, ένα κενό, ένα χάσμα που έχει εντοπίσει το σύστημά μας, πολύ ενισχυτικό. Ελπίζω ότι τις κατάλαβα τις ερωτήσεις Την έκθεση κανένα σχόλιο. Περιμένουμε ακόμα. Οι επενδυτές στην Banco Popular περιμένουν. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τίποτε παραπάνω, απλώς να μεταφέρουμε στην... Στην Deloitte ότι Είμαστε σε φάση νόμιμης αναμονής. Για τη Λεπτονική Τράπεζα, αυτό που πρέπει να βεβαιώσουμε είναι ότι η εθνική νομοθεσία περί πτωχεύσεων ισχύει και εφαρμόζεται και ότι θα είναι το αποτέλεσμα με άλλων κατώμελων σε περιπτώσεις πτώχευσης. Δεν ξέρω αν καλά κατάλαβα την ερώτησή σας. Αυτό δεν είχε να κάνει με το έντις. την εγγύηση των καταθέσεων. Σε κράτη-μέλη που έχουν περισσότερες από μία διαδικασίες περιπτωχεύσεις ε, υπάρχουν ίσως περισσότερες δυνατότητες. Έχουμε 19 και διαφορετικέ διαδικασίες στοχεύσεων και διαμοτεύσει σχετικά με το ΕΝΤΙΣ. Ε, Δικαίω έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθεια να σπρώξει τη συζήτηση με την ιδέα στην πρώτη φάση της συζήτησης να υπάρχει ένα σύστημα αμοιβαίας δανειοδότησης, δηλαδή όχι χρήση, του κινδυνού, αλλά μόνο μια δυνατότητα χρηματοδότησης Συμμετέχουμε στην τεχνική δουλειά για το ΕΝΤΙΣ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν είμαι σε θέση να πω τι θα γίνει και αν θα υπάρξει αντίκτυπο στο σύστημα, στο σύστημα τα σχόλιά μου ήταν ότι μακροπρόθεσμα θα ήταν πολύ καλό να γίνει ένα σύστημα διάθεσης εξυγένωσης της Ευρωζώνης. Αλλά για να υπάρξει αυτή η επικέντρωση στο ευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να υπάρξει και ένα δίκτυο ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις καταθέσεις. Πολύ γενικό το σχόλιο. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, μάλιστα. να και πάλι. είστε ναι, στο catch Ήταν χρόνο ομιλία των ε, ομάδων. Δεν θέλετε. Ο κύριος ορτασούν. Ευχαριστώ κύριε Κένικ. Πολύ γρήγορα. Από τα λόγια σας καταλαβαίνω ότι θα θέλατε το εργαλείο να το έχετε και στη φάση πρώτης εξυγένσης. Την συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη και στην περίπτωση της Banco Popular θεωρούμε ότι έχουμε το πρόβλημα της ε, υποβάθμισης των ε, ρευστών στοιχείων. Η άλλη ερώτησή μου όμως έχει να κάνει με το κενό στο καταστατικό που μπορούν να ζητήσουν οι αρχές από, τις τα υποκείμενα παράγωγα. Ε, δεν ε, ισχύει αυτό προς στιγμήν. Είναι ένα κενό στο καταστατικό και θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε. Ποια έποψή σας. Ναι, δεν θα σχολιάσω για το μορατόριο πάλι, απλώς για τα MRL πάντοτε ζητούσαμε ελαστικότητα, ιδίως για τα υποκείμενα MRL. Είναι μια απόφαση της τράπεζας, ειδική του τραπεζικού τομέα, οπότε δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με το κενό στο καταστατικό. Αλλά αν έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ύψος, ελπίζω θα μπορούμε παντότε να μείνουμε σε ένα... και ευχαριστώ. Κύριε Κένιγκ, θα ήθελα να επανέλθω στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, όπου αναφέρονται πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων ότι το Συμβούλιο σας είναι ακόμα στην φάση της ε, σύστασης και χρειάζεται κατανόηση. Το ερώτημα όμως είναι ποιες ε, είναι οι προτεραιότητες σας και με κατάπληξη διάβασα στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου πως δεν ήταν σε θέση ε, να ορίσει και να ονομάσει τις κρίσιμες λειτουργίες της τράπεζας, όλων των τραπεζών που εποπτεύει το Συμβουλίο σας. Ε, νομίζω ότι αυτό θα ήταν πρώτη προτεραιότητα. Έτσι, γιατί εσείς συντονίζετε τα Μπέιλιν και μόνο εσείς ε, αξιολογείτε την ε, συστημική σημασία της κάθε τράπεζας. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω. Για ποιον λόγο δεν είστε σε θέση να ορίσετε τις κρίσιμες λειτουργίες των τραπεζών που εποπτεύετε. Η δεύτερη μου ερώτηση το ελεγκτικό συνέδριο επίσης ε, λέει ότι καταλήξατε στην εκτίμηση ότι δεν έχει εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Οδηγία Εγγύησης των Καταθέσεων ε, και δεν θα είναι όλες οι χώρες σε θέση να σώσουν μια μεγάλη τράπεζα ή να εγγυηθούν τις καταθέσεις εάν καταρρεύσει. Είδου λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ως νομοθέτες. Μπορείτε σας παρακαλώ να κατονομάσετε σε ποιες χώρες κατά την εκτίμησή σας δεν έχει εφαρμοστεί η οδηγία. Ε, είδατε στο πρόσωπό μου ότι ε, απόρρισα κάπως με τη δεύτερη ερώτησή σας. Θα πρέπει να ξαναδώ την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά για να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση, το ελεγκτικό συνέδριο στην αξιολόγησή του, στο, έκανε την αξιολόγησή του τέλος του 16, αρχές του 17. Τότε ακόμα εξετάζαμε εξέτασε το ελεγκτικό συνέδριο όπως είπε ακριβώς ε, το τι κάναμε και τότε ακριβώς χαρτογραφούσαμε τις κρίσιμες λειτουργίες των τραπεζών και αξιολογήσαμε τώρα ακριβώς τις κρίσιμες λειτουργίες σε κάθε μία τράπεζα αλλά ο συνήθως επειδή ε, ο τραπεζικός τομέας είναι περίπλοκος, έχουμε ακόμα κάποια ερωτηματικά, όπου λέμε εντάξει μπορεί να είναι κάτι το κρίσιμο αυτό, αλλά θα πρέπει να το ξαναδούμε το 18. Οπότε είναι μια διαδικασία, το 16 πράγματι ίσχυε αυτό. Δεν είχαμε χαρτογραφήσει όλες τις ε, κρίσιμες ε, λειτουργίες. Το 17 υπήρχε ένα αστείο στον διάλογο με τον ε, κλάδο, γιατί λέγαμε ότι ζητώντας την αυτοαξιολόγηση είχαμε πολύ μεγάλες τράπεζες οι οποίες κατέληξαν στο ότι είχαν δύο-τρεις λειτουργίες που ίσως ήταν κρίσιμες και πολύ μικρές τράπεζες είχαν 50 ε, εξαιρετικά ε, κρίσιμες λειτουργίες. Οπότε υπάρχει πολύ διαφορετική εμπειρία στην κάθε τράπεζα και τώρα ήδη το 17 τα εναρμονίσαμε αυτά, το τι είναι δηλαδή κρίσιμες λειτουργίες, ε, το τι ε, μπορεί να αντικατασταθεί και ότι μόνο δεν αντικαθίσταται εύκολα ακριβώς μας απασχολεί. Οπότε θα έλεγα ότι τα ευρήματα εκεί του ελεγκτικού συνεδρίου το 2016 έχουν αντιμετωπιστεί, αλλά οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει περαιτέρω. Δεν είναι λοιπόν θέμα λάθος προτεραιοτήτων. Πρώτη προτεραιότητα το 2016 ήταν ακριβώς να έχουμε μια εικόνα τι εικόνα έχουν οι τραπεζικοί όμιλοι και ποιες ήταν οι προτεραιότητές μας. Τώρα, εγώ αντιλαμβάνομαι, αλλά ίσω κάνω όλα. Συγγνώμη, όχι, δεν μιλάω για το έντις, μιλάω για την οδηγία. Ναι, ναι, τα συστήματα εγγύηση καταθέσεων έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη, όσων γνωρίζω. Το σύστημα εγγύηση των καταθέσεων έχει αποκλήσει. αποκλήσεις, κάποια κράτη-μέλη έχουν ενσωματώσει το περίφημο άρθρο 11, το δικαίωμα μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού. άλλε ε, το έκαναν μέσω Paybox, αλλά εδώ πέρα ειλικρινά πρέπει να ξαναδιαβάσω έκθεση του συνεδρίου, γιατί εγώ είχα καταλάβει κάτι διαφορετικό, ότι έχουμε σύστημα εγγύηση των καταθέσεων και το να ελέγχουμε την σωστή εφαρμογή της οδηγίας είναι αποστολή της ε, Κομισιόν. Εάν εμείς συνειδητοποιήσουμε κάποιο έλλειμμα θα ειδοποιούσαμε την Κομισιόν και θα λέγαμε αυτό βρήκαμε, φροντίστε το και επιληφθείτε. Ε, α, μπορείτε επίσης ε, να απαντήσετε και γραπτός ε, τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ολοκληρώνουμε λοιπόν. Είχαμε μία επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και σας ευχαριστώ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 We take both offense that they didn't even warrant it. So, dear colleagues, we need to we move to the next point. Um, which is the last. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι και το τελευταίο. Κοινό σύστημα ΦΠΑ, υποχρέωση ελάχιστο κοινού συντελεστή. Ορίστηκα εγώ εισηγητής από το Προεδρείο και επειδή είναι πολύ απλό το θέμα, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε βάσει του, ε, του άρθρου 15, απλουστευμένη διαδικασία. Το σχέδιο κειμένου έχει ήδη διανεμηθεί και λίγη σε δύο μέρες η προθεσμία για την ε, υποβολή ένστασης ή αντίρρησης. Εάν δεν προβάλλει αντίρρηση ένσταση η αντιρρηση εαν δεν προβαλλει αντιρρηση εστω και ενα μέλο τη επιτροπή, θα θεωρηθει εγκεκριμενη η εκθεση χωρί τροπολογίε και θα πάει απευθεία στην Ολομέλεια. Τι αφορά η έκθεση. Είναι διαδικασία διαβούλευση, άρθρο 113 της συνθήκης και είναι μια μικρή αλλά σημαντική συνιστόσα του συνόλου συστήματο για το ΦΠΑ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όπω γνωρίζετε, έχει πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες, όμως αυτό το συγκεκριμένο τμήμα ουσιαστικά καθορίζει ως μόνιμο χαρακτηριστικό τον ελάχιστο κοινό συντελεστή 15% για τον κλασικό ΦΠΑ και που ισχύει όπως συμφωνήθηκε το 92. Και έκτοτε έχει λάβει συστηματικά πολλές παρατάσεις για να συνεχίσει να ισχύει. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το μετατρέψει σε μόνιμο συντελεστή, δεν είναι και κάτι επαναστατικό, διότι είναι κάτω του κλασικού συντελεστή που είναι 17%. Και συμφωνώ ότι 15% είναι καλό ποσοστό, άρα καλωσορίζω την μετατροπή του συντελεστή σε μόνιμο. Η έκθεση Απλώς εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χωρίς περαιτέρω σχόλια. Καλό τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν και να ανιγνωρίσουν το νομικό κενό στο πρόγραμμα δράσης του ΦΠΑ και όπως ξέρετε ε, είναι σημαντικές οι υπόλοιπες διατάξεις αλλά όχι στην έκθεση αυτή το κάνεις σε αυτήν την ε, συζήτηση δεν μας ενδιαφέρουν αυτά ακόμα. Θετική αποτίμηση λοιπόν της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κάνει μόνιμο τον ελάχιστο κοινό συντελεστή του 15%. Δεν βλέπω τους σκιώδης μου, αλλά βλέπω τον κύριο Ζήλε. Κύριε Ζήλε παρακαλώ, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ εκ μέρου ε, του κυρίου Σάντρι Λούνε, επειδή εκείνο ήταν σκιώδη εισηγητή από του συντηρητικού μεταρρυθμιστέ. Να πω ότι ο κύριο Λούν απλώ θέλει να θυμίσει ότι το 1992 έχει δώσει παράταση 6 φορέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό συμφωνούμε απολύτω με αυτήν την έκθεση διαβούλευση, η οποία προβλέπει το σύστημα αυτό σε μόνιμη βάση. Ώστε το 15% να εφαρμόζεται ως ελάχιστος κοινό συντελεστής. Ε, γιατί όπως ξέρετε τα κράτη-μέλη μας εφαρμόζουν ε, προς στιγμή 17% συνήθως. Άρα το 15% δεν είναι πρόβλημα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλα σχόλια, Περφάνσου πρόεδρε και εισηγητή. Ευχαριστούμε για την πρόταση αυτή που πιστεύω μόφωνα θα εγκριθεί. Απλώς είναι ευκαιρία να πούμε ότι για τους ελάχιστους κοινούς συντελεστέ χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να ενοποιηθεί κάποια στιγμή. Σωστά λοιπόν είπατε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί αντικείμενο συνένεσης και είναι και κάπως βιαστικό το θέμα. Διότι έχει εγκριθεί το πακέτο ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να γίνει αυτό σύντομα για να περάσουμε από το μεταβατικό σύστημα. Το να εγκρίνουμε τον ελάχιστο κοινό συντελεστή ε, ως ένα μέρος αυτής της διαδικασίας δεν μας λύνει το κάθε πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλος κανείς συνάδελφος να ζητά το λόγο. Όπως ξέρετε, οι προθεσμία για την ε, υποβολή ένστασης ή αντίρρησης είναι σε δύο μέρες. Μόλις εκπνεύσει στις 23 Μαρτίου η προθεσμία αυτή, θα πάμε απευθείας στην Ολομέλεια στην 1η του Απριλίου. Ευχαριστώ. Κυρίσουμε τη λήξη της συνεδρίασης αυτής. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα την Δευτέρα 26 στις 3 και 3η πρωί. Να σας θυμίσω ότι αύριο στις 2.30 θα έχουμε εργαστήρι κοινό με την Επιτροπή ε, Προπολογισμών για την δημοσιονομική δυνατότητα της Ευρωζώνης. Να θυμίσω ότι όσοι συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας για την Τραπεζική Ένωση και τα MPL αύριο θα υποφεληθούν. και με τον κύριο Αρτουή επίσης θα τα δούμε αυτά, ενώ έχουμε επιτροπή τη Δευτέρα. Ευχαριστώ. Λίγη συνεδρία.